Καλημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Μαριά για τις ε,